εδώ στο Κοινοβούλιο και να απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων του. Δεύτερη ανακοίνωση από το ΕΛΚ και τους σοσιαλδημοκράτες. Ο πρόεδρος δέχτηκε αλλαγές στις επιτροπές και οι διορισμοί αυτοί θα γίνουν σήμερα. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις στη στιγμή